Alors, je pense qu'on va commencer. Euh, donc, on est au point 7, euh, droit de l'homme. Ah. Αρχίζουμε, λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε με την ε, ευρωπαϊκή πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο του 2018. Έχουμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης που έγινε ήδη τον Οκτώβριο και που παρουσιάζει τι συνολικέ τάσει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και τι δυσκολίε. Και βάσει των συμπερασμάτων τη ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Ένωση, διατυπώνονται συστάσει για να δούμε πώ θα διατυπωθεί μια πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθούνται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Θα συζητήσουμε σήμερα τι τροπολογίε στην έκθεση αυτή. Έχουν υποβληθεί 487 τροπολογίες που υπάρχουν στο πρωτότυπο και στα αγγλικά. Η Επιτροπή Γυναικών για τα Δικαιώματα της Γυναίκας έχει υποβάλει γνωμοδότηση υπό τη μορφή επιστολής που θέλουν να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Η ΑΦΕΤ θα συνεδριάσει στις 4 συνεδρίου για να ψηφίσει την έκθεση αυτή. Η έκθεση αυτή στη συνέχεια θα υποβληθεί στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Η ετήσια έκθεση τη Επιτροπή Εξωτερικών Προποθέσεων για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια θα εγκριθεί και αυτή στην Ολομέλεια. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ιζαμπέλ Βίσλερ, η οποία θα μας ενημερώσει για την γνωμοδότησή της και για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί σε αυτή και να δούμε ποιες θα μπορέσουν να σωματωθούν στην έκθεση. Παρακαλώ. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τις 487 τροπολογίες που βάλατε. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις που να είναι για όλους ικανοποιητικέ. Ωστόσο, θα πρέπει να όλοι να έχουμε κατά νου ότι προκειμένου να παραμείνει εύληπτη η έκθεσή μας, να μην παραμένει και σχετικά συνοπτική. Πολλές τροπολογίες αφορούν τις ηθαγενείς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους υπερασπιστές τους και τις διάφορες μειονότητες. Θα προσπαθήσω να ε, καταρτήσω νέες συμβαστικές λύσεις για τα θέματα αυτά. Κάποιες τροπολογίες σκοπό είχα να έχουμε νέους υποτίτλους για κάποια θέματα. Θα ήμουν λίγο επιφυλακτική εδώ Ας προσπαθήσουμε να μην κατονομάσουμε κάποιους, αλλά να δώσουμε την ίδια έμφαση σε όλες τις ομάδες ε, πληθυσμών και μειονότητες. Νομίζω οι τροπολογίες 47, 185 κτλ. είναι τέτοια παραδείγματα. Ωστόσο υπάρχουν πολλές τροπολογίες μεταξύ άλλων για τους ΛΟΑΔ, οι οποίες θα ε, συμπεριληφθούν οπωσδήποτε στις συμβαστικές λύσεις Λίγες τροπολογίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένε αναφορές σε χώρες. Οι 170, οι 246, οι 270, 271, οι 331 και 332. Όπως είπαμε, είναι ευαίσθητη η περίπτωση να κατονομάζουμε συγκεκριμένε χώρε και έτσι κινδυνεύουμε να παραμελήσουμε κάποιε. Θα έλεγα λοιπόν να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώ, χωρί να μιλάμε για συγκεκριμένε χώρε και να προσθέσουμε στα παραρτήματα, σε δύο παραρτήματα, τα καταπήγοντα ψηφίσματα που έχουμε ε, ε, υπόψη για συγκεκριμένε χώρε και συγκεκριμένε περιπτώσει. Να υπάρξει δηλαδή η αναφορά των χωρών αυτών στα παραρτήματα. Μιλάμε για τρίτε χώρε. Γι' αυτό η τροπολογία 101 που αναφέρει ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνεται. Οι τροπολογίες 130 και 131 το ίδιο και κάποιες άλλες. Για την 187 που μιλά για την αναβάθμιση της Επιτροπής μας σε τακτική επιτροπή, ακόμη και αν η ιδέα πολύ μου αρέσει, πιστεύω ότι δεν είναι το σωστό σημείο για να επιληθεί ένα τέτοιο θέμα και θα πρέπει να γίνει μια ευρεία συζήτηση μεταξύ όλων μόνο. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, έχουμε πολλές τροπολογίες οι οποίες θα συμπεριληφθούν στις συμβαστικέ λύσεις προκειμένου να υποβάλουμε συστάσεις και να καλύψουμε, ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη δυσκολία και αλλαγή. Η τροπολογία 371 μου αρέσει πολύ γιατί μιλάει για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού ε, διεθνώς. Ένα πολύ σημαντικό ε, σκέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να το προσέξουμε. Προκειμένου να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Οι υπεύθυνοι ε, εγκλημάτων πολέμου και γενοτοκτονιών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπερίληψη ε, τροπολογιών για την ατιμορρησία. Ανέφερα την τροπολογία 253, 54 και 55. Ε, μου είχατε πει και την προηγούμενη φορά ότι είχα μακρηγορήσει, γι' αυτό θα κλείσω εδώ την παρέμβασή μου και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όταν δούμε με λεπτομέρειες τις επιμέρους τροπολογίες. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλ. Έχουμε σοβαρή έλλειψη ε, σκιωδών εισηγητών και εισηγητριών. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θέλουν να λάβουν το λόγο εκ μέρου του κυρίου ε, Κόσελιν που δεν είναι εδώ. Μαρία. Ε, ε, Ευχαριστώ Μαρία. Ευχαριστώ την Ισαβέλ για τη δουλειά της. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες, αλλά φυσιολογικό. Ενδιαφέρει πολύ συνήθως το Κοινοβούλιο το θέμα αυτό και ο καθένας θέλει να δώσει τη δική του άποψη για αυτό το σημαντικό θέμα. Ως ομάδα Έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες για τα θέματα ΛΟΑΔ. Θεωρούμε ότι δεν τονίζεται αρκετά. Θέλουμε να τονιστεί περισσότερο στην έκθεση το θέμα αυτό. Επίσης και για τα δικαιώματα των γυναικών. Και για τις αντιπροσωπίες. Κατά τα άλλα, η έκθεση αυτή θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσελκύσει πολύ περισσότερο την προσοχή του σώματος και ευχαριστούμε την Ισαβέλ και ελπίζουμε η εργασία της ε, να είναι αντικείμενο προσοχής από τις άλλες ομάδες, όπως από τη δική μας. Ευχαριστώ. Για την ομάδα ΡΙΝΙΟΥ, τον Σαρλ Γκέρενς, θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Η κυρία Ροντρίγεθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την καταπληκτική εργασία που έκανε η συγκήτριά μας, την συγκήτρια δηλαδή για την καταπληκτική εργασία της. Υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες με βάση και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών. Όπως είδαμε χθε στην Επιτροπή μας, κάποιοι φορείς συγγνώμη, κάποιες ομάδες του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα ε, ευάλωτες και κυρίως ε, η κοινότητα των ΛΟΑΔΚΙ υφίσταται πολλές διακρίσεις σε πολλά μέρη του κόσμου. Και τώρα, η κατάσταση των γυναικών στον κόσμο, όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν επαρκεί. Θέλουμε να τονίσουμε πολύ περισσότερο πόσο πολλές είναι οι περιπτώσεις ε, βίας κατά των γυναικών. Και επίσης, υπάρχουν πολλές ε, άθλιες πρακτικές κατά της σωματικής ακαιρεότητας των γυναικών για παράδειγμα, η γενετήσια, η γενετήσιοι και η ε, καταναγκαστική γάμη σε πολύ μικρή ηλικία. Μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες, υφίστανται πολλά προβλήματα. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της εμπορίας γυναικών. Επίσης, κάποιες τροπολογίες θέλουν να τονίσουν την ε, μείωση της βιοπικιλότητας ε, λόγω της κλιματικής αλλαγής ε, που έχει επιπτώσεις και για τους ανθρώπους φυσικά. Δεν είναι μόνο ότι ορισμένοι αρνούνται καν την κλιματική αλλαγή, αλλά κάποιες επιχειρήσεις έχουν άθλιες πρακτικές που καταστρέφουν τους βιοτόπους και καταστρέφουν γενικότερα το περιβάλλον και δεν επιτρέπουν να ζει κανείς αξιοπρεπώς. Και νομίζουμε ότι η σύνδεση της, ε, των προβλημάτων της βιοπικιλότητας με τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να τονιστεί περισσότερο στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πράσινους κανείς. ECR, ουδής. Γκουε, ουδής. Οπότε, οι συνάδελφοι, εάν θέλω να πάρω τον λόγο. Α, Παρακαλώ, Ισαβέλ. Απλώς να τονίσω τη σημασία της έκθεσης αυτής και την όλη συζήτηση που γίνεται σχετικά. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την άριστη δουλειά της, διότι είναι μια πολύ καλή αφετηρία για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Προφανώς υπάρχουν πολλές προτάσεις τροπολογιών και εμείς από πλευράς μας υποβάλαμε πληθώρα. Ελπίζουμε λοιπόν με το διάλογο που θα οργανώσουμε μεταξύ μας θα μπορέσουμε κάπως να τις ε, σκεφτούμε και να διευρύνουμε το φάσμα του πεδίου της εκτρίου αυτής γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις γυναίκες, με τις μειονότητες, με την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών την καταπολέμηση της βίας ε, εις βάρος των γυναικών, το θέμα των ηθαγενών, θέματα που θα θέλαμε να καλύπτονται από την έκθεση και να αναφερθούν ρητός και ελπίζουμε ότι η συγγήτρια θα δείξει αρκετή διαλεκτικότητα για να αποδεχτεί τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ Ιζαμπέλ. Θα δώσω το λόγο στην Τζεπελβής τώρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έχει γίνει για την έκθεση αυτή, γιατί έχει να κάνει και με τις σχέσεις του Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά τα προγράμματα δράσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω οι συστάσεις μας να είναι συστάσεις που θα συμπεριληφθούν και στο έργο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, εξωτερικής δράσης. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω από βάθους καρδιάς πραγματικά να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο. Γιατί όταν βλέπουμε πόσες πολλές τροπολογίες έχουν ε, υποβληθεί, καταλαβαίνουμε το ενδιαφέρον του κόσμου και τη δουλειά που έχει γίνει από πίσω. Ευχαριστώ και τη γραμματεία βέβαια της Επιτροπής μας και τη γραμματεία της ομάδας μας και στις δικές μου υπηρεσίες του γραφείου μου, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο που έχει κρατήσει πολύ και έχουν συμμετέχει πολύ σε αυτό. Θα ήταν πραγματικά κρίμα. Αναφέρθηκε Δεκεμβρίου, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βλέπετε ότι οι σκιώδες δεν είναι, και ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για συνεδριάσεις δεν φτάνει. Έχουμε και το Στρασβούργο, οπότε μήπως μπορούμε να αλλάξουμε την ημερομηνία για να μην ε, κάνουμε μια δουλειά μετά από όλα όσα έχουμε όλοι προσφέρει, να μην καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις ιδέες που έχουν διατυπωθεί θα έπρεπε μη τι άλλο να έχουμε να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε τις συναντήσεις που χρειάζεται για να καταλήξουμε σε σεβασμούς που θα ικανοποιούν όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Πέρασε το μήνυμα στους κοιόδους εισηγητές νομίζω για να φροντίσουν να είναι διαθέσιμοι για να προχωρήσει η δουλειά γιατί οι προθεσμίες είναι προθεσμίες. Όσο πιο αργά είναι έτοιμη η έκθεσή μα, τόσο λιγότερο θα ληφθεί υπόψη από τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Και θα ήταν κρίμα. Οπότε το μήνυμα περνάει νομίζω στις πολιτικές ομάδες και τους σκιώδες εισηγητέ ώστε να φροντίσουν να βρουν το χρόνο για να διατυπωθούν οι συμβαστικέ τροπολογίε. Τώρα, δυστυχώ πρέπει να διακόψουμε. Δυστυχώ, ευτυχώ, τέλο πάντων, θα έχετε τη δυνατότητα να πάτε για καφέ. Γιατί το σημείο 8 που είναι μετά, θα, για αυτό το σημείο στις παρατέταρτο παραδέκα θα έχουμε τους ε, ομιλητές μας γι' αυτό. Οπότε σταματάμε για ένα τέταρτο 20 λεπτά.